Dear colleagues, let's now move to... Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία για τα benchmarks. Και επιτέλους λοιπόν ψηφίζουμε για το θέμα αυτό, τους δείκτες αναφοράς, είχαμε αναβολές ε, διάφορες και τώρα επιτέλους περνάμε στην ψηφοφορία. Είμαστε μόνο στα πλαίσια της εικόνα. Κάνουμε καινούργια λοιπόν δοκιμαστική ψηφοφορία. Πέρας. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε. Τροπολογία 26. NV1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Με προφορική τροπολογία της ΑΛΔΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Στη σελίδα 8. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 104. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. πέρας. Απορρίπτεται η ισοψηφία. Μήπως Μπράια να κάτσετε εκεί για να σας βλέπω καλύτερα. Μάλιστα. 109. Και η επόμενη. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνοντα. 111. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 111. Ψηφίζουμε. Πέτερ, έχετε την κάρτα σας. Την έχετε την κάρτα σας. Πολύ ωραία. Πέρασε. Εγκρίνεται, κοιτάξτε. Πάλι καλά που το ελέγξαμε. Ευχαριστώ πολύ και θα λάβω υπόψη τη νέα ε, ισοζυγία, αν θέλετε. Πάμε λοιπόν στην 10, 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 100. Έλεγχο, έλεγχο. Εσεί είχατε σημειώσει υπέρ, μάλιστα. έλεγχο, έλεγχο λοιπόν για την 113. Εκατόν δεκατρία. Ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 114. Έλεγχος παρακαλώ γιατί είναι λίγο περίεργες οι ισορροπίες. Πέρας. ισοψηφία απορρίπτεται. NV20 υπέρ. Κατά. Ε, έλεγχος για το NV20. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 21 κατά. Είναι ψήφι. 115 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 115. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 20 κατά. Συμβαστική β' υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 145 και 146 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 159. Υπέρ. Σοσιαλιστές είναι υπέρ. Έλεγχος παρακαλώ για την 159. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 19 υπέρ. 16. Κατά. Ψηφίζουμε παρακαλώ έλεγχο για την 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε ή με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Έλεγχος, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεμβιβαστική ε. Τροπολογία 29 λοιπόν. Τροπολογία 29 στη σελίδα 18. Μακάρθη. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κα... και 2 υπέρ κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 και NV3 υπέρ, κατά. Η πράσινη είναι κατά, απορρίπτεται. 34 και NV4 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά. Έλεγχος για την 4 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρασε. 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά πίπτων, 36 λοιπόν. Διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Έλεγχος για την 36. Έλεγχος. Για την 36 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Καταπίπτει. 39. Και unblock ε, τα ιδεολογικές σκέψεις. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται. Σε μη η 42 μάλλον και NV8, υπέρ. Έλεγχος, ηλεκτρονικός, ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 43, υπέρ. Κατά. Έλεγχος, παρακαλώ, για την 43. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-21. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ Έλεγχος, παρακαλώ, για την 74 ψηφίζουμε. Πέρασε. 22 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική μη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. σειράς. 42 ψήφοι υπέρ, μία κατά, 0 αποχές. Ψηφίζουμε την απόφαση έναρξης των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων με ονομαστική κλίση και πάλι έναρξη ψηφοφορίας. Έχουμε ακόμα κάποιου συναδέλφους που δεν έχουν ψηφίσει. Μάλιστα, πέρασε. 39 ψήφοι υπέρ, μία κατά, Έχουμε λοιπόν ειδική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη συνεδρίαση. 10 Ιανουαρίου στι 9 το πρωί η επόμενη συνεδρίαση. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Ξεκουραστείτε και να περάσετε καλά στις διακοπές.